Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση και θα τα πω από εδώ και πέρα ουγγρικά. Λοιπόν, Καταρχάς, να δούμε το πρώτο σημείο της διάταξης, έγκριση μερίσιας διάταξης. Ενημερώσαμε την Τετάρτη όλες και όλους σας και αναφέραμε την έκθεση για την για το θεματολόγιο 2020 ήταν ένα σημείο το οποίο αναβλήθηκε για αργότερα. Συμφωνείτε με τη μισή διάταξη όσοι έχει τοποποιηθεί συμφωνείτε. Δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών. Έχετε στο φακελό σας τα πρακτικά. Υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά. 14-15 Μαρτίου. Αν όχι, προτείνω να θεωρήσουμε τα πρακτικά εγκεκριμένα αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Τρίτο σημείο, ανακοινώσεις της Προέδρου. Διερμηνία. Έχουμε τις εξής γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, δανικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εστονικά, ουγγρικά, λιφανικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά, ρουμανικά. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η σημερινή μας συνεδρίαση και τώρα 14 Μαρτίου 2016 έχουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουν αποσταλεί σε όλους τους βουλευτές τα πρακτικά τη συνεδρίαση των συντονιστών 16 Μαρτίου θεωρούμε ότι εγκρίνονται αποφάσεις αυτές εφόσον δεν αντέδρασε κανείς και δεν παραπονέθηκε κανείς σε σχέση με αυτές τις αποφάσεις. Ολοκληρώνω λοιπόν εδώ και τις ανακοινώσεις Προέδρου. Έχουμε μια νομοδότηση που θα πρέπει να ψηφίσουμε. Είπα ότι η έκθεση Κρασνοντέψκη για τη... Το θεματολόγιο 2020 αναβλήθηκε. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία τη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τη σήμανση των μεθόδων για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στι καταληκτικέ παρατηρήσει κτλ. Η Επιτροπή Απασχόληση είναι καθήλυνα αρμόδια. Η συγγήτρια είναι πρόεδρο Σιλβία Κώστα, που δυστυχώ δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. 25 Φεβρουαρίου έληξε η προθεσμία για τις τροπολογίες. Κατατέθηκαν 71 τον αριθμό τροπολογίες. Περνάμε στην ψηφοφορία. Έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Kezdhetjük. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Okay, and uh, switch uh, to English if it's better. Αν καλύτερα να τα πω αγγλικά από εδώ και πέρα. Συμβιβαστική ένα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουν ηλεκτρονικά έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται πράγματι. Τροπολογία 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2, ψήφι περ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25, ψήφι περ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4, ψήφι πέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32, ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7, ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8, ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39, ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, άλλο θα ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Έχουμε μια προφορική τροπολογία από τον Γιώχαν Κιουκτσουκ. Ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46, ψήφι πέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11, ψήφι πέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 67 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73 ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Νομίζω. θα το ελέγξουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προπολογία 75. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογία 76. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Ψήφι ΠΕΡ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 ψηφιπέρ. κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, άρχεται ψηφοφορία. Okay. If anybody will... Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Σα ευχαριστώ συνάδελφοι. Yes. Το αποτέλεσμα είναι 25 υπέρ, 0 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Να συνεχίσουμε τώρα με τα υπόλοιπα σημεία. Σιωπή παρακαλώ. Συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε. Επόμενο σημείο. στρατηγική η Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2014-2020 και την χάνει να είμαι εγώ η εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο ενέκριναν αυτή τη στρατηγική και αυτή είναι η δική μας απόκριση, η έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας. Η πολιτική μας ε, για την νεολαία είναι πολύ σημαντική για να καταλάβουμε τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι νέοι. Γνωμοδοτήσεις επέβαλαν και άλλες επιτροπές, η Επιτροπή ΕΜΠΛ και ΚΟΝΤ, η Επιτροπή δηλαδή Ελέγχου των Προπολογισμών και η Επιτροπή Επασχόλησης και τοποθετήθηκαν για τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τον Δεκέμβριο οργανώσαμε στις 13 του περασμένου μήνα μια σημαντική συνεδρίαση για την στρατηγική περνεολαία. Ήταν ε, παρόν και ο αρμόδιος επίτροπος και το όλο θέμα συζητήθηκε κατά λεπτός. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 25 Απριλίου στις 3 το απόγευμα. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 30 Μαΐου. Και ως εισηγήτρια θα ήθελα να παρουσιάσω τα βασικά σημεία της έκθεσής μου. Ως εισηγήτρια λοιπόν πρέπει να πω ότι αυτό είναι ο τρίτο κύκλο τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για του Νέου και αποτιμούμε τους, ε, κατά πόσο επιτύχαμε του στόχου που είχαμε θέσει ως τώρα. Το ανθρώπινο κοινωνικό κεφάλαιο που εκπροσωπούν οι νέοι είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενεργητικού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθοριστικά για το μέλλον μα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και για τα κράτη-μέλη. Πρέπει γι' αυτό να αξιοποιήσουμε στο το δυνατόν περισσότερο το δυναμικό αυτό προ τη δημιουργικότητα, τι δεξιότητε των νέων γιατί η οικονομική κρίση έχει πλήξει κατεξοχήν τους νέους και τις δυνατότητες απασχόλησής τους. Ορισμένοι έχουν ε, εξοφηθεί στην περιθωριοποίηση της, ε, από την κοινωνία και η, η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ε, από το γεγονό ότι κάποιοι από του νέου περιθωριοποιούνται, αποκλείονται από την κοινωνία και πολλέ φορέ οδηγούνται και σε βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Γι' αυτό το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε τι προσπάθειές τη για να βελτιώσει την απασχολησιμότητα και την ένταξη των νέων στην αγορά απασχόληση, την κοινωνική του ένταξη και την ενεργό του συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα πρέπει να βρούμε λύσεις σε σημαντικά προβλήματα όπως την καταπολέμηση τη ενεργείας, της ενεργείας των νέων όλους ιδιαίτερως, την βελτίωση της, του βιωτικού του επίπεδου και των ε, προοπτικών του για το μέλλον, την κοινωνική του ένταξη και την καταπολέμηση της βίαιης ρίζοσπαστικοποίησης. Αυτή είναι η βασική μα στόχη. Για την επιδίωξή του χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ε, θεσμικών οργάνων, των Ευρωπαϊκών Κρατών, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των λοιπόν Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Χρειάζεται μια συντονισμένη προσέγγιση και ολοκληρωμένε πολιτικέ λύσει για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τι κοινωνικέ πολιτικέ, την πολιτική απασχόληση, την πολιτιστική πολιτική, τον αθλητισμό και την υγεία. Αυτή είναι η βασική τομή δράση. Το επόμενο διάστημα προγραμματισμού μεταξύ 2016-2018 θα πρέπει ενεργώς να προωθήσουμε τη συμμετοχή των νέων σε διάφορους τομείς δράσης που θα τους βοηθήσουν να βρουν δουλειές και να γίνουν ενεργοί πολίτες. Ο εθελοντισμός, η ενεργό συμμετοχή στην, ε, στα πολιτικά πράγματα προωθούνται μέσω του προγράμματος Εράσμους εν μέρη και τα κοινωνικά ταμεία, καθώς και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τους Νέους, ε, παίζουν σημαντικό ρόλο. Εάν δούμε τι γινόταν στο προηγούμενο διάστημα προγραμματισμού, βλέπουμε ότι υπήρχαν έτσι καλλιώς θετικές τάσεις, Πρέπει λοιπόν να το σημειώσουμε αυτό, αλλά πρέπει σίγουρα να δίνουμε και τις προσπάθειές μας. Μπορούμε ακόμη να κάνουμε πολλά. Παραμένουν ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, οπότε πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε προβλήματα όπως η εγκατάλειψη του σχολείου σε πρώιμες ηλικίε. παρόλο που εδώ υπάρχει μια τάση βελτίωσης, ο αριθμός των νέων που ολοκληρώνουν την ανώτερη εκπαίδευση αυξάνεται, αλλά παρόλα αυτά, στην ηλικιακή ομάδα 20-24, όλο και περισσότεροι, τελειώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όμως τα 20 έως τα 24 κάποιοι όλο και περισσότεροι φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η συμμετοχή των νέων στον πολιτικό βίο με τα κοινωνικά μέσα, τα μέσα δικτύωσης ε, είναι ο κατεξοχήν τρόπος που χρησιμοποιούν και θα πρέπει να παρακολουθούμε και αυτήν τους, ε, την συνήθεια για την εμπλοκή του στα πολιτικά πράγματα. Το ίντερνετ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το 2014 κάθε νέος, ένας στους δύο νέους ήταν μέλος κάποιου συλλόγου και ένας στους τέσσερις είχε κάποια εθελοντική δράση. Αυτό επίσης είναι πολύ θετικό και πρέπει να βελτιωθεί, να ενισχυθεί η τάση αυτή. Το να βρίσκεται ποιοτική θέση εργασίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για πολλούς νέους γιατί τους καθυστερεί η μία έβρεση εργασίας από το να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια και να γίνουν γονεί. Η απασχόληση των νέων μειώνεται. Οι αριθμοί μας ε, ανησυχούν. 1,7 εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη είναι άνεργοι ή αναζητούν εργασία. Πάνω από 3 εκατομμύρια νέοι δεν έχουν εργασία, ούτε, κατά, ούτε ασχολούνται με κατάρτιση ή εκπαίδευση και βεβαίω εκπαιδευση και βεβαιώς η φτωχεια και ο κοινωνικό αποκλεισμός είναι μια απειλή για 27 εκατομμύρια νέους. Το ποσοστό ένδυας για τους νέους είναι μεγαλύτερο από ό,τι για τους πιο ηλικιωμένους και αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Η μερικού χρόνου εργασία και η μακροχρόνια ανεργία είναι χαρακτηριστικές τάσεις για τους νέους της Ευρώπης. Η περιθωριοποίηση παρουσιάζεται και εκδηλώνεται διαφορετικά μεταξύ των διαφορετικών ομάδων νέων. Αυτοί που προέρχονται από οικογένειες φτωχότερες, από οικογένειες μεταναστών, ή ανήκουν σε κάποια είδου μειονότητα που έχουν δηλαδή δυσκολότερες ε, συνθήκες ή που μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε κάποιο ε, ορφανοτροφείο ή με γονιούς που έχουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο ε, ξεκινούν τη ζωή τους με τεράστιο μειονέκτημα δεν προχωρούν προς την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση. Επίσης αυτή που έρχονται από άλλε οικογένειε αυτοί που μπορούν να ταξιδέψουν, που ενθαρρύνονται να σπουδάσουν και να καλλιεργηθούν, έχουν πολύ περισσότερε ευκαιρίε και έχουν πολύ λιγότερε πιθανότητε να γίνουν περιθωριοποιημένοι ή να ριζοσπαστικοποιηθούν. Η έκθεσή μου αποτελείται από τέσσερα βασικά κεφάλαια. Το πρώτο είναι οι γενικές συστάσεις, το δεύτερο η απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, το πρωτο ειναι οι γενικέ συστασεις το δευτερο η απασχοληση εκπαιδευση και καταρτιση το τριτο ο ρόλος της χρηματοδότησης και το τέταρτο η συμμετοχή στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αυτά είναι τα τέσσερα σημαντικότερα κεφάλαια στα οποία έχω επικεντρωθεί και στο πρώτο, στις γενικές συστάσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε διορθωμένο διάλογο με τους νέους, με τις οργανώσεις νέων και να έχουμε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό ε, σύστημα συνεργασίας για τις πολιτικές για τους νέους συνδυάζοντας όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα. Πρέπει κυρίως να στραφούμε σε οργανώσεις σε περιφερειακό επίπεδο που μπορούν πραγματικά να δώσουν μορφή στην ε, πολιτική των νέων, στις ε, ενώσεις των οικογενειών, την εκκλησία που μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Κεφάλαιο 2, στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. Το όπως υπόθηκε χθες και στην κοινή, στην κοινή συνάντηση με τις επιτροπές Κόντ και ΕΜΠΛ, είναι σημαντικό να στραφούμε στις δεξιότητες, τα λεγόμενα skills. Χρειάζεται καλύτερος συντονισμός, διότι η αγορά εργασίας μεταλλάσσεται. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η συνεργασία μεταξύ των φορέων της αγοράς εργασίας και των εκπαιδευτικών είναι σημαντική, διότι διαφορετικά δεν θα έχουν οι νέοι τις δεξιότητες που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας και δεν θα βρίσκουν και δουλειά. Στην ε, επίσημη και άτυπη αλλά και την διαβίου μάθηση είναι πολύ σημαντικό τι δεξιότητες ε, θα διδάξουμε στους νέους. Η αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων επίσης και των προσόντων είναι σημαντική. Η διασυνοριακή αναγνώριση εννοώ είναι ουσιαστική σημασία σε αυτό για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Επίσης, κάνω λόγο για το πρόγραμμα Erasmus ε, συν και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αλλά τώρα να περάσω στο κεφάλαιο 3. Οικονομική πόρη, χρηματοδότηση. Ε, στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να αναφέρουμε το Erasmus συν την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, τα κοινωνικά ταμεία, την εγγύηση για τους νέους και τα διαστατικά ταμεία, τα ταμεία μάλλον συνοχή, συγγνώμη. Μπορούν όλα αυτά να βελτιώσουν την καλύτερη ένταξη των νέων στην αγορά εργασία στην Ευρώπη. Βεβαίω, χρειάζονται και νέε πρωτοβουλίε και νέα προγράμματα. Στο κεφάλαιο 4 τώρα, για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και τη συμμετοχή των νέων σε αυτήν. Εδώ τονίζω τη σημασία τη ε, συμμετοχή των νέων σε αυτή τη διαδικασία διότι θέλουμε να αποφασίζουμε για αυτούς αλλά μαζί τους. Επίσης τονίζω τη σημασία του αθλητισμού και των κοινωνικών δραστηριοτήτων, αλλά ταυτόχρονα τη σημασία της εθελοντικής εργασίας. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της εκθεσής μου. αλλά επειδή υπάρχουν αυστηρά όρια για τον αριθμό χαρακτήρων που μπορεί κανεί να συμπεριλάβει στην εκθεσή του, αναγκαστικά περιορίστηκα σε κάποια σημαντικότερα θέματα. Γι' αυτό θα υποβάλω και περισσότερε τροπολογίε για να επιμηκύνω το κείμενο. Αν υπομονούμε να ακούσουμε τι αντιδράσει σα, τι αντιδράσει των σκιωδών εισηγητών, αλλά και των μελών τη Επιτροπή μα. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Και τώρα Έχουμε περίπου 30 λεπτά στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Να ξεκινήσουμε με τους Σκιώδης και μετά με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Μπορείτε να μας κάνετε νόημα αν θέλετε το λόγο. Οι σκιώδεις θα έχουν 2-3 λεπτά και οι υπόλοιποι 1-2. Πρώτος, η πρώτη, Ο κύριος Νέκοβ. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ απόλυτα με όσα υπόθηκαν μόλις. Επίσης ως προς τις τροπολογίες μου Ας αρχίσω με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, 57% των οργανώσεων νέων πιστεύουν πως η οπτική τους γωνία δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη κατά το σχεδιασμό πολιτικών για τη νεολαία. Πιστεύω πως η φωνή των οργανώσεων της νεολαίας πρέπει να ακούγεται κατά τη χάραξη πολιτικών λόγω της εμπειρογνωμοσύμινης και της εμπειρίας τους. Τα στοιχεία και οι εκθέσεις δείχνουν πως οι νέοι έχουν ιδιαίτερα μειονεκτήματα, ειδικότερα οι λεγόμενοι ΝΕΤ. Είναι οι νέοι οι οποίοι δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση, κατάρτιση ή εργασία. Οι μετανάστες επίσης έχουν μειονεκτήματα. Γι' αυτό και η πιο αποτελεσματική δράση που μπορούμε να αναλάβουμε πρέπει να προσανατολίζεται στην απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων όπως είναι επιχειρηματικότητα και η μεγαλύτερη κινητικότητα. Αυτά μπορούν να ενθαρρύνουν τους νέους να έρθουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, μπορούμε να τους κοιμάσουμε καλύτερα για τη μελλοντική του ζωή. Πέραν αυτού, πιστεύω πως ο αθελοντισμός πρέπει να ενισχυθεί. Στη χώρα μου, τη Βουλγαρία, εργάζομαι ενεργά για την πρόθεση του εθελοντισμού εδώ και δύο χρόνια. Υπό το πρίσμα της προσφυγικής κρίσης πιστεύω πως η εθελοντική εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα εξωτερικά μας σύνορα όπως και στα κέντρα υποδοχής και καταγραφής. Οι νέοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο, σε εθελοντική εργασία πρέπει να αναγνωρίζονται πως συμμετέχουν σε μία μορφή άτυπης κατάρτισης. Η στρατηγική αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε μορφές άτυπης εκπαίδευσης. Θα μας δώσει επίσης, θα δώσει επίσης ευκαιρίες στους μετανάστες να αποκτήσουν ένα πτυχίο και μια θέση εργασίας, καθώς άνθρωποι με μια θέση εργασίας δεν είναι πλέον πρόσφυγες. Έτσι δίνουμε ευκαιρίες τόσο στους μετανάστες όσο και στους νέους. Επόμενος, ο κύριος Σάντης, ζήτησε το λόγο. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει. Κύριε Χοντή. Ε, δεν άκουσα καλά. Νομίζω ότι δώσατε το λόγο σε μένα. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, για να μην χάνουμε χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάβασα την ανακοίνωση της ε, Κομισιόν για τη Στρατηγική για την Νεολαία, διάβασα και την έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά επειδή είναι και σύντομο ο χρόνος, αναρωτιόμουν αν αυτά που λέει η Κομισιόν, η δική σας έκθεση νομίζω ότι είναι, κάνει μια προσπάθεια να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, αλλά θα έλεγα ε, κάποιες παρατηρήσεις δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα σήμερα που ζει η νεολαία της Ευρώπης. Θα έλεγα λοιπόν, αν αυτά που γράφουμε μέσα στα κείμενα και εμείς με μεγαλύτερη ευθύνη γιατί είμαστε αιρετοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πηγαίναμε και τα λέγαμε στους νέους της πατρίδας μου εγώ είμαι από την Ελλάδα. Αλλά βγάλτε την Ελλάδα, πείτε η κατάσταση κτλ. Σε αυτού του νέου που ξενυχτάνε στι πλατείε τη Γαλλία και στο Παρίσι για τα αιτήματά του. Τι θα μα λέγατε. Ούτε οι διαπιστώσει μα είναι ακριβεί, αγαπητοί συνάδελφοι, και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί για την νεολαία έχουμε όλη ευθύνη, ανεξάρτητα από πολιτικέ τοποθετήσει και ιδεολογικέ, έχουμε σε ευθύνη. Τιμάζουμε χαμένε γενιέ, Τι τους υποσχόμεθα τι προσπάθειες κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Έχω λοιπόν την εντύπωση πως δεν αποτυπώνεται σωστά η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η νεολαία και οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί, το ποσοστό της ανεργίας των νέων, το ποσοστό των νέων που είναι κάτω από το όριο της στόχιας και μεγάλα ποσοστά που δεν έχει καμία ελπίδα για μια ένα καλύτερο ποιοτικό επίπεδο καθώς έχει ανασφάλεια για την απασχόλησή του. Το κάνουμε ανταγωνιστικό βλέποντας τους άλλους ως εχθρούς σε μια κοινωνία που της λείπει η συνοχή και η ευαισθησία απέναντι στα προβλήματα της νεολαίας. Και γίνεται αυτό αγαπητοί συνάδελφοι διότι οι πολιτικές που ακολουθούνται οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθούνται δεν μπορώ να μην το χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο τα είδαμε και χθε στην κουβέντα οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα. Αν δηλαδή την εκπαίδευση την αποδώσεις στους νόμους και στις δυνάμεις της αγοράς δεν θα έχει αυτό που εσύ ζητά για να διαμορφώσει ανθρώπου, ενεργού πολίτε ή για να δημιουργήσει τι προποθέσει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Δεν θέλω να σα κουράζω περισσότερο, διότι συνήθω σε τέτοιε εκθέσει βρίσκομαι σε αυτό το δίλημα. Εντάξει, να κάνουμε κάποιε προσπάθειες. Είμαστε όμω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε εκλεγμένοι. Πρέπει τουλάχιστον να αποτυπώνουμε τα προβλήματα Α πούμε, στι διαστάσει που υπάρχουν. Δεν λέω πω ε, η συγγήτρια δεν έχει τέτοια πρόθεση. Ε, η προσπάθειά τη είναι πιο συγκεκριμένη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι με αυτέ τι στρατηγικέ δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη νεολαία τουλάχιστον κατά τι διακηρύξει. Βεβαίω θα έχουμε νέου ημιμαθεί με υλική κατάρτιση, ανασφαλή όσο αφορά το χρόνο, και τις συνθήκες εργασίας, ανταγωνιστική όσο αφορά τους άλλους νέους, χωρίς καμιά κοινωνική αλληλεγγύη, να προσπαθήσουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτή τη ζούγκλα. Θα έχουμε και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Αλλά δεν θα έχουμε όμως μια γενιά στην οποία μπορεί να ελπίζει ο ευρωπαϊκός λαός και η ευρωπαϊκή λαή σε κάτι καλύτερο ως ένα συλλογικό όραμα για μια καλύτερη κοινωνία. Ε, να σταματήσω εδώ, θα κάνω και τις επιμέρους παρατηρήσεις, Κατά τα άλλα θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι εκτιμώ την προσπάθεια, τη φιλότιμη προσπάθεια της συγγήτριας, αλλά <laughs> τα γεγονότα και η εικόνα νομίζω πως είναι ας πούμε, πιο, πιο δραματική. Ευχαριστώ πολύ που μου ακούσατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συνάδελφοι. Κυρία Μποτσκούρ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανέγνωσα την έκθεσή σας και πρέπει να σας συγχαρώ για το εξαιρετικό της περιεχόμενο και για την ε, οπτική γωνία που έχετε υιοθετήσει. Συμφωνώ με πάρα πολλά σημεία, αλλά σε κάποια θα πρέπει να δοθεί, πιστεύω, μεγαλύτερη έμφαση και να ενισχυθούν. Λόγου χάρη είναι πολύ σημαντικό η ιδέε και η φωνή των ενώσεων και των συλλογών νέων να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζουμε πολιτικές για τους νέους. Οι ενώσει τη νεολαίας είναι καθοριστικές για την επιτυχία αυτή τη. στρατηγικής. Στην έκθεσή σα, δίνεται έμφαση στη σημασία των ε, ομάδων νέων και στα πλαίσια του διορθωμένου διαλόγου μεταξύ ε, των νέων και των πολιτικών ενθυνόντων. Θα πρέπει να τονίσουμε επίσης την ε, απόκληση που υπάρχει μεταξύ των προσόντων και των δεξιοτήτων που διδάσκονται στου νέου και τι ανάγκε τη αγορά εργασία. Αυτό το έχει εντοπίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να εργαστούμε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δεν μπορούμε παρά να ενισχύουμε τα κράτη-μέλη στο να ασχοληθούμε με το πρόβλημα αυτό. Είναι καθοριστική σημασία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να χρησιμοποιηθεί με πιο αποτελεσματικό και στοχευμένο τρόπο. Τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα θα πρέπει να απλουστευθούν για να μπορούν να είναι και εύχρηστα. Πολλέ πτυχέ δεν μπορούμε να τι λεχθούμε ωστόσο ω πολιτική ομάδα λόγου χάρη την περισσότερη χρηματοδότηση προς τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν πώς να ε, οργανώνουν τις δαπάνες τους. Οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν πραγματικά μεγάλα προβλήματα. Πολλοί από αυτούς ε, έχουν απογοητευτεί πλήρως. Πρέπει λοιπόν να ε, επενδύσουμε και στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας ταυτόχρονα. Δεν γνωρίζω εάν ε, μπορώ να κλείσω αισιόδοξα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την ε, ευημερία, για την ε, αισιόδοξη πρόπτικη για τους νέους μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Κύριος Μαραγκάλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπόσκορ. Εγώ νομίζω ότι θεωρώντας δεδομένο ότι αυτά που λέγονται στην έκθεση δεν μπορούν παρά να μας βρουν σύμφωνους, είναι αποδεκτά όσο ορθά και συνεκτικά όσα περιγράφεται στην έκθεσή σας. Βέβαια και σε άλλες εκθέσεις της Επιτροπής μας έχουμε πει και ξαναπεί τα ίδια. Ε, νομίζω ότι έχουμε όλη επίγνωση ε, του ότι πολλές φορές έχουμε πει και γράψει τα ίδια ε, τον τελευταίο χρόνο στην Επιτροπή μας. Πρέπει όμως να γίνει αυτή η συζήτηση και πρέπει να υποθούν και να γραφτούν αυτά που είπατε. Να προσθέσω τώρα κάποιες δικές μου σκέψεις. Νομίζω ότι ίσως ξεχνάμε το γεγονός ότι αυτό που συμβαίνει στη νεολαία μας αντικατοπτρίζει και αυτό το οποίο γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και γενικότερα. Δηλαδή η νεολαία δέχεται τι επιπτώσει των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, των ε, πολιτικών ε, πρόνοια, ευημερία, ε, πλήττεται από τι περικοπέ, τη λιτότητα, τι περιστολέ των δημοσίων δαπανών σε διάφορε χώρε κτλ. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισορροπίες στην πρόσφατη κοινή ευρωπαϊκή ιστορία Άρα βλέπουμε νομίζω και τις επιπτώσεις ε, του πώς εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική και της μη γης κάποιων ε, πολιτικών προσαρμογής, διαφορετικών πολιτικών κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο εντός του οποίου τελικά οι νέοι μας ε, και με κάποιες διαφοροποίησεις αλλά και με πολλά κοινά χαρακτηριστικά ε, έχουν όλες αυτές αρνητικές επιπτώσεις να υποστούν. Είπα ότι υπάρχουν τα χαρακτηριστικά κάθε χώρα, παραγωγικά μοντέλα, οικογενειακή τυπολογία, αστικά μοντέλα κτλ. κτλ. Όλοι αυτοί οι παράγοντε συνεισφέρουν. Αν όμως ε, μπορούμε να δώσουμε μια γενική κατεύθυνση τι να πούμε, αλλάξτε πολιτικές και αλλάζουν και οι επιπτώσεις. Ε, σίγουρα αυτό είναι μια λύση, αλλά πρέπει να δούμε και τα αίτια και τις επιπτώσεις. Εγώ θα έλεγα δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, το έγγραφο, όπως είναι λογικό, καταγράφει αυτό που υπόθηκε και πριν, ότι δηλαδή είμαστε σε ένα πλαίσιο που την αρμοδιότητα την έχουν τα κράτη-μέλη, εντάξει, συμφωνούμε από αυτού. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να έχει ένα ρόλο συντονιστή, ε, να προσφέρει καθοδήγηση, προσανατολισμό, υποστήριξη. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να ζητήσουμε και από εμάς τους ίδιους αλλά και από την Κομισιόν είναι πέραν αυτού του ρόλου για το συγκεκριμένο ζήτημα να έχει ένα ηγετικό ρόλο, να δώσει όθηση να βοηθήσει να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή ε, στις πολιτικές αυτές, ε, όχι με κοντόθωρο τρόπο, ομοιόμορφο, αλλά να γίνεται σεβαστή και η αρμοδιότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν αποφάσει. Πάντω η Κομισιόν θα πρέπει να διατυπώσει προτάσει για μια πραγματική αλλαγή και πάντα ανάλογα με την κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Δεν ξέρω αν μπορεί η Κομισιόν να προτείνει κάποια κοινά πλαίσια δράση, αν μπορεί να υπάρχουν επίση κάποια πλαίσια ενό μόνιμου benchmark, να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά δίκτυα. Καλά σχεδιασμένα. Είναι μια άλλη πρόταση για να δούμε τι κάνουν οι άλλοι και να το εφαρμόσουμε και εμείς βέβαια κατά το δοκούν. Και τελικά πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, κάποιους δείκτες ε, για τον προσδιορισμό προτύπων κτλ. Δεν είναι κάτι εύκολο βέβαια σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας ρόλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να ολοκληρώσω. Κάτι που λέγεται στην έκθεση, είναι προφανές, αλλά πρέπει να επιμείνουμε. Είναι ότι πρέπει τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, την Νεολαία και άλλα προγράμματα, θα πρέπει να τα ε, εναρμονίσουμε κατά κάποιο τρόπο για να πετύχουμε συνέργειες. Διότι αν δεν το πετύχουμε αυτό υποπίπτουμε για μια ακόμη φορά στο σφάλμα ότι ε, ρίχνουμε ε, λεφτά στα προβλήματα, όπως λέγεται. Είναι ίσως ε, κάπως γραφικό αυτό σαν εικόνα, αλλά περί αυτού πρόκειται. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την κοινή, τη μεικτή αποτελεσματικότητα και τη διαδικτύωση, τη διασύνδεση των προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά δε, το European Youth Initiative, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Νεολαία, είναι ένα καλό στοιχείο, αλλά ο προεπολογισμό έχει παγώσει. Διότι δεν ξέρουμε ακόμα πώ θα τον αξιοποιήσουμε και περιμένουμε και από την Επιτροπή Προπολογισμού τη σχετική εκτίμηση. Δεν έχουμε ακόμη όμω κάτι στα χέρια μα. Αυτή η έκθεση λοιπόν θα μπορούσε και θα έπρεπε την άποψή μου να ασκήσει κάποια πυρός προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή θα πρέπει να ε, πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε κύριος ο κύριος Χουντής αν τα είχα πει εγώ δεν θα τα είχα πει τόσο καλά είμαι βέβαια γι' αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διάφορες χώρες, αναφερθήκαμε χθες ε, στην Πολωνία. Για παράδειγμα, όπου οι νέοι πολύ πιο εύκολα μπορούν να, να βρουν απασχόληση σε κάποια επιχείρηση σε σχέση με άλλες χώρες. Πρέπει να ξέρετε, δεν έχουμε όλοι τους ίδιους κανόνες. Στην Γαλλία, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και από διοικητικής πλευράς ε, να προχωρήσει κανεί σε ίδρυση μια επιχείρηση και από οικονομική πλευρά υπάρχουν δυσκολίε. Υπάρχει λοιπόν ε, δουλειά που μπορεί μπορεί να γίνει και από κοινού αλλά και ξεχωριστά σε κάθε χώρα γιατί δεν υπάρχει ισότητα. Αν θέλετε να μας το λύσω ό,τι αφορά την εργασία. Ευχαριστώ. Κυρία Φερχάιεν. Δύο πράγματα σε σχέση με τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να ανοίγουν σχολεία σε κάποιες χώρες, σε κάποιους τομείς είναι λίγο μια κλειστή υπόθεση. Η ανάληψη επαφών δεν θεωρείται κάτι θετικό, αν και αυτό χρειάζεται για να μπορέσουν οι μαθητές να πάνε μπροστά μπροστά. Πιστεύω πως χρειαζόμαστε μια άλλη κουλτούρα ως προς το μοντέλο αυτό για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τώρα το να νομίζουμε πως μόνο μέσω επιχειρηματικότητα και προσόντων των νέων μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων πιστεύω ότι είναι λίγο αφελές. Αφετέρου πρέπει να δούμε πως και για αυτούς οι οποίοι δεν αποκτούν τα προσόντα τους, αυτούς που εγκαταλείπουν το σχολείο, για τους νέους οι οποίοι δεν έχουν κάποια επαγγελματική κατάρτιση, ότι για όλους αυτούς πρέπει να αναπτύξουμε εναλλακτικά μοντέλα για το πώς με άλλον τρόπο μπορούν να αποκτήσουν προσόντα. Και πιστεύω εδώ μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον για μοντέλα ορθότερων πρακτικών όπως αυτά υπάρχουν σε άλλες χώρες και πως πρέπει να σκεφτούμε πως η ένα προς ένα εφαρμογή είναι δύσκολη επειδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά στο πλαίσιο των στρατηγικών για την νεολαία πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να μετεμφυτεύσουμε τέτοια παραδείγματα σε άλλα συστήματα και εδώ μπορούμε να συνοδεύσουμε αντίστοιχα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί μια ορθή πρακτική σε ένα άλλο σύστημα ή πώς πρέπει να τρομοποιηθεί και πιστεύω πως απομένουν πολλά να κάνουμε στον τομέα αυτό για να δημιουργήσουμε προοπτικές για νέους οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλές, υψηλά προσόντα αλλά ταλέντα και ικανότητες η μη τυπική εκπαίδευση παίζει σε αυτό το πλαίσιο ένα σημαντικό ρόλο κατά την απόψή μου. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αποκλειστικά από τον τυπικό τομέα της εκπαίδευσης, αλλά πρέπει να δούμε πώς ικανότητες, βασικά προσόντα, ικανότητες που χρειάζεται να έχει κανείς για να επιβιώσει στην αγορά εργασίας, πώς μπορούμε να τα φέρουμε αυτά στους νέους, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν έως τότε, και δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα κατεστημένα συστήματα. Γι' αυτό και πρέπει να σκεφτούμε για εναλλακτικά μοντέλα και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που παίρνω το λόγο τώρα. Δεν δηλαδή θα ήθελα να συνεχίσω αυτό που είπε η προλαλήσασα θα σκεφτούμε τι χρειάζονται οι νέοι. Πρώτα απ' όλα χρειάζονται μια καλή εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση που θα τους προετοιμάσει να γίνουν ενεργοί όχι μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά επίσης στη ζωή τους. Και δεύτερον, στην αγορά εργασίας χρειαζόμαστε σαφείς μηχανισμούς, οι οποίοι θα προωθούν την απασχολησιμότητα και την απασχόληση της νεολαίας, των νέων. Όσον αφορά την εκπαίδευση, έχουμε έναν τυπικό στόχο εντός της στρατηγικής μας Ευρώπη 2020. Αφενός θέλουμε να μειώσουμε το ποσοστό αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο ή την κατάρτιση προώρα και το δεύτερο να αυξήσουμε το μερίδιο των ανθρώπων με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αφέτερου η αγορά εργασίας και αυτό που προσφέρει δεν ανταποκρίνεται στους στόχους μας. Στην ομάδα αυτή έχουμε έναν μεγάλο αριθμό νέων οι οποίοι είναι απλά απογοητευμένοι. επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλο το δυναμικό τους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και πιστεύω πως πρέπει να προωθήσουμε την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση περισσότερο από ποτέ σε διαφορετικά επίπεδα. Επειδή εκεί μπορούμε να βρούμε πολλές προσφορές θέσεων εργασίας. Το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Στη διαδικασία της εκπαίδευσης σημαντικά είναι τα διδακτέα προγράμματα. Σε διαβούλευση με επιχειρήσεις πρέπει να καταρτίζονται με τις προσδοκίες της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, χρειαζόμαστε επίσης ομαδική εργασία σε διάφορα προγράμματα δεν γίνεται διδασκαλία της ομαδικής εργασίας. Η επιχειρηματικότητα είναι σημαντική, αλλά η επιχειρηματικότητα καθ' αυτή δεν θα τα λύσει όλα. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, πρέπει να προωθήσουμε και να ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε να προσλάβουν νέους. Ίσως κάποιες φοροαπαλλαγές επί ένα ή δύο χρόνια θα τους ενθαρρύνουν να προσλάβουν νέους. Ή μια συγχρηματοδότηση των εξόδων εργασίας, του κόστους εργασίας. Η ανταλλαγή πρακτικών είναι πολύ σημαντική σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό που μου λείπει από την έκθεση, η οποία είναι πολύ καλή και την οποία εκτιμώ πολύ, αυτό που μου λείπει ωστόσο είναι μια αναφορά στο γεγονός πως πρέπει να προωθήσουμε πρωτοβουλίες όπως το Γιούρις. Την μαθητεία, την εργασία, έτσι ώστε οι νέοι να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες να μπορούν να βρουν, πού μπορούν να βρουν θέσει εργασία. Είναι ένα στοιχείο στη ζωή των νέων το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το ζήτημα τη στέγη και τη πρόσβαση σε στέγη. α μην το ξεχνούμε. Οι νέοι, εάν πάρουν μια θέση εργασία εάν θέλουν να εργαστούν, χρειάζονται στέγη. Χρειάζεται να μείνουν κάπου. Είναι ένα βασικό αγαθό, μια βασική ανάγκη. Και αυτό μου λείπει στην έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ με την έκθεση και πιστεύω και εγώ αυτό που λέτε εδώ, ότι δηλαδή υπάρχει ανάγκη πιο συστηματικής συνεργασίας ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για την νεολαία. Και σε ό,τι αφορά στο πού τοποθετείται οι, πολιτικοί, πολιτικές για τη ε, νεολαία και αν ακούγεται και πόσο η φωνή των νέων. Ε, με απογοήτευσε πολύ ε, στη διακοινοβουλευτική συνάντηση που είχαμε πριν τα Χριστούγεννα το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της δικής μου κυβέρνησης ούτε καν ήρθε για να μιλήσει σε αυτή τη συνάντηση. Έδειξαν ε, μία έρευνα που είχε γίνει μεταξύ λίγων κρατών μελών που για μένα κατέδειξε σημαντικές ελλείψεις ε, και της δικής μου κυβέρνηση ό,τι αφορά την πολιτική για την νεολαία και για την παιδεία και μίλαγαν μόνο για στόχους, για δακτέα ύλη, πραγματικά μια πάρα πολύ κοντόθωρη άποψη για την παιδεία. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν πολλές ε, πολιτικές ε, και μέθοδοι μάθησης ε, δασκαλίας που μπορεί να είναι πολύ θετικά παραδείγματα προς μίμηση από τα κράτη-μέλη και νομίζω ότι έχουμε πολλά να διδαχθούμε από τον άλλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επισφαλή απασχόληση, ένα σύντομο σχόλιο, οι νέοι συχνά πέφτουν θύμα εκμετάλλευσης αδίστακτων εργοδοτών. Τα μέτρα λιτότητας είχαν ως αποτέλεσμα όλο ε, και περισσότερες συμβάσεις ε, ε, με πολύ, από πολύ αδίστακτους εργοδότες που εκμεταλλεύουν τα παραθυράκια της νομοθεσίας και επιβάλλουν πολύ αρνητικούς όρους στους νέους που τελικά και τα είπατε και εσείς για τη στέγαση για παράδειγμα δεν θέλουν, ένα δεν θέλουν μια αξιοπρεπή κατοικία. Οι νέοι δεν θέλουν να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή στο μέλλον, να φτιάξουν οικογένειε κτλ. Είναι πολύ δύσκολο όμω ε, να σκεφτούν οτιδήποτε άλλο όταν δεν γνωρίζουν ούτε καν κατά πόσον θα έχουν ένα μισθό στο τέλο τη εβδομάδας ε, και εθελοντισμό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάποιε οργανώσει, ε, κάποιε χώρε, κάποιοι εργοδότε, κάποιε οργανώσει, χρησιμοποιούν τον εθελοντισμό ως ένα τρόπο για να εκμεταλλεύονται ακόμη περισσότερο τελικά τους νέους. Ε, δεν πρέπει να γίνεται έτσι, αλλά ο εθελοντισμός πρέπει να οδηγεί ε, σε κάτι άλλο, όχι να κάνεις κάτι για το τίποτε, αλλά να είναι ένας δρόμος προς την απασχόληση. Και ο εθελοντισμός δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει το κράτος. Εντάξει, καλό είναι ο εθελοντισμός να ενθαρρύνουμε τους νέους, αλλά να οδηγεί και κάπου αυτό. Επίσης, οι νέοι τελικά στις δομές εξουσίας και στους θεσμούς ε, βλέπουν ότι έχουν μια θέση, θεωρούν ότι εκπροσωπούνται τους χάρη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί αν δεν ε, βλέπουν κάτι τέτοιο χάνουν την ελπίδα τους. Γι' αυτό βγήκαν στους δρόμους στο Παρίσι, γι' αυτό έχουν, ε, το, έχουμε το κίνημα Occupy. Είδατε και τι έγινε και στα, το Σάββατο κατά των μέτρων λιτότητας. Αν δεν βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ και ιδίω αυτοί που θεωρούν ότι είναι διαφορετικοί, ή θεωρούν, παραδείγματο χάρη, όλοι αυτοί οι ΛΟΑΔΜ που θεωρούν ότι είναι διαφορετικοί, πώς, ε, που τοποθετούνται σε αυτή τη κλίμακα εξουσία, ε, άτομα με αναπηρία, ε, του άσυλο κτλ. Ε, νιώθουν αυτοί οι νέοι ότι λαμβάνονται υπόψη οι δικέ τους απόψεις και οι ανάγκες. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερη εμπλοκή και συνεργασία με τους νέους, αλλά με τους δικούς τους όρους και να βρούμε έναν τρόπο να τους φέρουμε πιο κοντά στα θεσμικά όργανα και να τους δώσουμε μια ισχυρή φωνή και όχι ε, να μείνουμε στα λόγια. Η έκθεσή σας, το δέχομαι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά και να ε, υποστηρίξουμε με πιο στεναρό τρόπο τους νέους και να τους δώσουμε ελπίδα. Ευχαριστούμε κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και νομίζω η έκθεση συμπεριλαμβάνει τα βασικότερα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Άλλωστε αντικατοπτρίζει και το διευθυμένο διάλογο που είχαμε με τους νέους. Δίνουμε έμφαση στην οικογένεια, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία και ούτω καθεξής. Και τον εθελοντισμό. Αυτά όλα αποτελούν μέρος των αξιών που συγκινούν τους νέους. Αν και πιστεύω ότι κάποιες πτυχές λείπουν εδώ, όπως οι επενδύσεις. Θέλουμε να επενδύσουμε στην ε, καλλιέργεια των νέων, δηλαδή να, καλλιεργήσουμε και στο, να επενδύσουμε και στο μέλλον της Ευρώπης. Πρέπει να βλέπουμε την ε, ενασχόλησή μας με τους νέους ως επένδυση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχουμε και κλήσει των οργανώσεων για τους νέους και τα παιδιά που ε, χρειάζονται χρηματοδότηση. Οι οργανώσεις αυτές αποτελούνται κυρίως από εθελοντές και όχι επαγγελματίες. Είναι λοιπόν δύσκολο να ε, χρησιμοποιεί κανείς περίπλοκα εργαλεία χρηματοδότηση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε στην έκθεση αυτή για να ευθυγραμμίσουμε τα, τα εργαλεία χρηματοδότηση που διαθέτουμε. Η κυρία Τρούπελ. Thank you. Yes, I would like to come back on a point we already discussed in our common here. Ευχαριστώ. Ε, μια, ένα θέμα που θέλω να ε, σχολιάσω γιατί τα είπαμε χθε και στην κοινή μας συνεδρίαση για την άτυπη εκπαίδευση. Έχουμε ήδη θίξει το θέμα αυτό και είναι πραγματικά σημαντικό να έχουμε μια ιδιαίτερη ματιά στους νέους που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Ότι ξέρουμε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτό είναι πρόβλημα και θα πρέπει ε, να δούμε τα αποδεικτικά στοιχεία που φτάνουν στα χέρια μας για τομείς όπως ο χορός, η το τραγούδι που έχουν πετύχει πάρα πολύ και έχουν επιτρέψει στους νέους να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα σχετικά προγράμματα και να καλλιεργήσουμε αυτές τις πρακτικές και να τις συμπεριλάβουμε στα στρατηγική μας. Διότι πολλοί είναι οι νέοι που έτσι ε, θέτουν τα θεμέλια για να προχωρήσουν μετά στην ανώτατη εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν να ε, κοιτάξουμε πολύ σοβαρότητα το πραγματικό νόημα της άτυπης εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Εάν με ενημερώνουν σωστά, εκ μέρους της Επιτροπής το λόγο θα πάρει ο κύριος Χαρτούν. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει το σχέδιο έκθεσης αυτό, καθώς στηρίζει και συμπληρώνει την προσέγγιση που επιλέξαμε για τη στρατηγική για τους νέους. Να τονίσω τρεις μεθόδους που θα έπρεπε να καλλιεργήσουμε περαιτέρω στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα, αυτό που σωστά αναφέρεται και στην έκθεση, στενή συνεργασία μεταξύ τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Πρέπει να συνδυαστούν και εφόσον συνδυαστούν σωστά, τότε μόνον μπορεί να επιφέρουμε αλλαγές. Το δεύτερο στοιχείο είναι η διατομεακή προσέγγιση. Η πολιτική για τους νέους, παρόλο που είναι, που είναι η αιχμή του δόρατος, δεν μπορεί να επιλύσει μόνη τη τα προβλήματα. Πρέπει να ε, συνδυάσουμε την απασχόληση, την εκπαίδευση και όλους τους σχετικούς τομείς. Και το τρίτο σημείο είναι να δώσουμε περισσότερο περιθώριο στους νέους ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν ακόμη τρία σημεία στα οποία θέλω να σταθώ. Πρώτον, ε, η σχέση μεταξύ απασχολησιμότητας και εκπαίδευσης. Το δεύτερο, πώς να καλύψουμε τις ανάγκες των νέων. Και το τρίτο, η συμμετοχή. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα. Πρέπει να δούμε την εκπαίδευση με έναν τρόπο πιο ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, θέλουμε οι νέοι να πετύχουν επαγγελματικά, κοινωνικά και στον ιδιωτικό του βίο. Ωστόσο, δεδομένου του υψηλού ποσοστού ανεργία, πρέπει να ε, δώσουμε έμφαση στην απασχολησιμότητα. Άρα, πρέπει να καλωσορίσουμε την ε, προσέγγιση σας στην έκθεση που δίνει έμφαση στην ε, εκπαίδευση μαζί με την επαγγελματική κατάρτιση. Επίσης, πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση τόνωσης της αποχειρηματικότητας, δηλαδή να επιτρέπουμε στους νέους να μπορούν να οργανώνουν όπως θέλουν τη ζωή τους. Και το τρίτο, το πιο σοβαρό στοιχείο μεταξύ όλων, είναι η αναγνώριση των δεξιοτήτων. Των δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι μέσω της άτυπης εκπαίδευσης. Το δεύτερο στοιχείο για τους νέους που δεν έχουν σχέση με την κατάρτιση, εκπαίδευση ή απασχόληση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μα, διότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο τέτοιων νέων μεγάλο αριθμό που δεν μειώνεται αρκετά. Οι ρυθμοί δεν είναι αρκετά αγοριά για να πούμε ότι, κάνουμε, ότι επιτελούμε πρόοδο. Χρειάζεται λοιπόν δράση σε συνεργασία με όλους τους τομείς. Και να υπογραμμίσω κάτι που είπαν και κάποιοι από τους ομιλητές. Δηλαδή η συνεργασία μεταξύ άτυπης και επισημης εκπαιδευση εκπαίδευσης. Πρέπει χέρι-χέρι να προχωρήσουν. Και τότε μόνο θα πετύχουμε σημαντική πρόοδο. Το δεύτερο υποστοιχείο αυτή τη προσέγγιση είναι να επικεντρωθούμε στη σωστή χρηματοδότηση, όχι μόνο με το πρόγραμμα Erasmus, αλλά και με τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία, τα Διευθυντικά και την ε, Πρωτοβουλία για του Νέου. Το τρίτο σημείο είναι η συμμετοχή. επιφανειακά φαίνεται οι νέοι να έχουν απογοητευτεί από τη ε, διαδικασία τη δημοκρατική και τα πολιτικά πράγματα. Αν όμω το εξετάσει κανεί προσεκτικά, θα καταλάβει ότι οι νέοι είναι πολύ ε, περίεργη. Ε, αυτό όμως το εξασκούν με τρόπους που δεν είναι συμβατή όσα σήμερα ισχύουν ε, ε, συνήθως. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε θέσει τρία επίπεδα γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα να ενισχύσουμε τον διαρθρωμένο διάλογο που να είναι και συστηματικός, να κοιτάξουμε τις προτεραιότητες των νέων για τη Νέα Ευρώπη και μετά να συνεχιστεί το πρόγραμμα Outreach, όπως ονομάστηκε, για τους νέους, με τα κοινωνικά δίκτυα και με, την, ε, με το συνδυασμό επιγραμμικών και μη επιγραμμικών μέσων, δηλαδή στο ίντερνετ. Τρίτο στοιχείο, Πρόεδρε. Η κρίση των προσφύγων έχει δείξει την δύναμη του εθελοντισμού, ιδίω των νέων στι κοινωνίε μα. Αυτό θα είναι ένα σημείο που πραγματικά θα ήθελα να ενισχυθεί και στο μέλλον, στη νέα στρατηγική, ε, την οποία θα αρχίσουμε τώρα να σχεδιάζουμε. Νομίζω ότι η έκθεσή σα θα είναι καθοριστική σημασία γι' αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρω, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν συνηθίζεται, αλλά θα παρακαλούσα μια ερώτηση στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, γιατί κάποιο πράγμα δεν το κατάλαβα. Είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι η συμπεριφορά της νεολαίας, αν το κατάλαβα καλά. Η πολιτική είναι κάπως ιδιόμορφη, ιδιότροπη. Αν το είπε έτσι, θα τον παρακαλούσα να το διευκρινίσει. Ευχαριστώ και πάλι. Ξέρω ότι δεν συνηθίζεται σε αυτή τη φάση διάλογος, αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα καταλαβαίνουμε καλά, μου φαίνεται. Κύριε Χουντή, ε, θέσατε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα του ξαναδώσω λοιπόν το λόγο του κυρίου Χάρτον για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση για τη συμπεριφορά των νέων. Παρακαλώ επαναλάβετε όμως την ερώτησή σας, διότι δεν άκουγε εκείνη τη στιγμή. Και πάλι συγγνώμη, διότι ξέρω ότι δεν συνηθίζεται, γι' αυτό ίσως και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν είχε τα ακουστικά του. Η ερώτησή μου είναι στο σημείο που είπε, ισχυρίστηκε ότι η συμπεριφορά της νεολαίας, η πολιτική συμπεριφορά, η κοινωνική συμπεριφορά της νεολαίας είναι κάπως ιδιόμορφη, είναι κάπως ιδιότροπη. Το κατάλαβα καλά. Αν το κατάλαβα καλά τότε μπορεί να μας πει δύο κουβέντες από πού βγαίνει αυτή η εκτίμηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε, με συγχωρείτε, την πρώτη φορά δεν ακούγα την ερώτηση. Αυτό που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις μας είναι ότι η συμμετοχή στις παραδοσιακές διόδους της πολιτικής ε, ζωής μειώνεται. Το βλέπετε από τη συμμετοχή των νέων στις εκλογές τοπικές, κοινοβουλευτικές ή ευρωπαϊκές το επίπεδο διαρκώ μειώνεται, ο αριθμό συμμετοχή. Από την άλλη όμω υπάρχουν κινήματα των νέων επιτόπου για πολιτικά προβλήματα, όπου πάρα πολύ γρήγορα μέσω των κοινωνικών δικτύων ενώνουν τις δυνάμεις τους, εκφράζουν τις απόψεις τους και τοποθετούνται ad για τα θέματα προκειμένου να έρθουν σε διάλογο με τους πολιτικούς ηθήνοντες και να τους πιέσουν να δράσουν. Από αυτό που είδαμε εμείς ως τώρα, από ε, τις ε, δυνάμεις των νέων που ενώνονται βραχυπρόθεσμα για ένα θέμα, ε, βλέπουμε ότι θέλουν να επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα και μπορεί να ξανασυνδυάσουν τις δυνάμεις τους για ένα επόμενο θέμα. Η προσέγγιση διαφέρει και ο τρόπος που χρησιμοποιούν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα είναι να το λάβουμε αυτό υπόψη για να τους δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες ώστε να ακούγεται τη φωνή τους και να λαμβάνεται υπόψη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω Μισολτάκη. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω, έλεγα λοιπόν, όλες και όλους ε, για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω και τους Κεώδης και όλους τους άλλους ε, βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού. Νομίζω ότι μπορούμε με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε να προσθέσουμε αυτές τις ιδέες που αναφέρατε εσείς σήμερα και να έχουμε έτσι μια πολύ καλή έκθεση. Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος ε, της έκθεσης, οπότε ίσως λόγω αυτών των περιορισμών να μην εστίασα όσο έπρεπε στις βέλτιστες πρακτικές και στο γεγονός ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διδαχθούν το ένα από το άλλο και να αξιοποιήσουν, να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ε, καλές πρακτικές για τις πολιτικές, τόσο για την νεολαία όσο και τις οικογενειακές πολιτικές. Πιστεύω λοιπόν ότι οι ιδέες σας, οι συστάσεις σας πραγματικά έχουν θέση σε αυτήν την έκθεση. Θα μπορούσαμε επίσης να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν θα μπορούσε περαιτέρω να βοηθήσει την νεολαία. Παραδείγματο χάρη, κάποιε φορά απαλλαγέ για τι επιχειρήσει που προσλαμβάνουν νέου ή κάποια οικογενειακά επιδόματα ή επίδομα στέγαση. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να στηρίξουμε την νεολαία και να βοηθήσουμε και όσους έρχονται από ένα κάπως πιο μειονεκτικό υπόβαθρο δεν ε, κατάγονται από μια πλούσια οικογένεια ή μπορεί να μην έχουν ένα πανεπιστημίου. Μπορούμε να του βοηθήσουμε λοιπόν ή την ε, εγκατάλειψη του σχολείου. Άτομα που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο προέρχονται από αδύναμα κοινωνικά στρώματα και αυτούς μπορούμε να τους βοηθήσουμε περισσότερο. Είπατε ότι έχει αλλάξει βασική ιδέα και θεωρία σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι θα πρέπει όλοι να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Αν όμως έχεις ένα μάστερ στις ε, καλές τέχνες για παράδειγμα δεν σημαίνει ότι θα βρεις και δουλειά στην αγορά εργασίας. Άρα είναι δύσκολο για τους νέους που μπορεί να έχουν ε, αποφυτίσει από ένα ανώτατο ε, ίδρυμα αλλά να μην βρίσκουν δουλειά. Μπορεί να μην χρειαζόμαστε χιλιάδες αποφύτους πανεπιστημίων ανωτάτων σχολών, αλλά χρειαζόμαστε ίσως άτομα που βγαίνουν από κάποια τεχνική σχολή και μπορούν να βοηθήσουν και στην αύξηση του ΕΠ της χώρας τους με τα τεχνικά τους προσόντα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη και τις παρατηρήσεις και ελπίζω ότι άπαξ και φτάσουμε στη συζήτηση των τροπολογιών θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε τροπολογίες συμβιβαστικές ε, που θα είναι αποδεκτές από τους περισσότερους και θα βελτιώσουν την έκθεση. Ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους για τις ε, υποδείξεις σας, για το έργο σας και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησιάς διάταξης. Να πω βέβαια κάτι που ξέχασα ότι 25 Απριλίου λίγη η προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών στις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο τη μερικέ διάταξη, που είναι η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και αύξηση τη πολυμορφία τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο μια ένωση κεφαλαίου αγορών. Συζητούμε λοιπόν ένα σχέδιο έκθεση. Αρμόδια καθήλυν επιτροπή είναι η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Εμεί συντάσσουμε γνωμοδότηση και ο συντάξης γνωμοδότηση είναι ο κύριο Λουίτσι Μοργάνο. Ξέρουμε ότι ΜΜΕ έχουν σημαντικό ρόλο στην ενιαία αγορά και η χρηματοδότησή του, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι κάτι που μα απασχολεί εδώ και καιρό. Υπάρχουν διαφορετικέ ε, κατηγορίε ΜΜΕ στα διάφορα κράτη-μέλη με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, οικονομικέ δομέ, ε, ανάπτυξη διαφόρων φάσεων κτλ. Η ΜΜΕ είναι επίση παρούσε και στι δημιουργικέ βιομηχανίε. Αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε προκλήσει. Ο κ. Μοργάνο παρατήρησε και ανέλησε αυτέ τι προκλήσει. Πριν δώσω το λόγο στον συντάκτη, στον ομοδότη, να πω ότι οι τροπολογίε θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι τι 25 Απριλίου στι 4 το μεσημέρι και η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα το Μάιο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά να μπορώ να υποβάλω στους ε, συναδελφούς αυτό το σχέδιο έκθεσης. Έχουμε να κάνουμε με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση των διαφορών της ποικιλομορφίας της χρηματοδότησης των ε, μικρομεσαίων και την πρόσβασή τους στις κεφαλαίες Μου φαίνεται σημαντικό ευθύς εξ αρχής να επισημάνουμε ότι πρόκειται για μία έκθεση πολύ στοχευμένα, κοιτάζει να προλάβει κάποια συγκεκριμένα σημεία που θα τα κοιτάξουμε σε μια κοινή επιτροπή για τις ε, σε μια κοινή έκθεση με την Επιτροπή ΙΤΡΕ που θα έχει τίτλο «Δημιουργική πολιτική χρηματοδότησης». Εδώ λοιπόν η έκθεση αυτή έχει πολύ στοχευμένη προσέγγιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να της δώσουμε λιγότερη προσοχή. Είναι λοιπόν σημαντικό ε, να ε, ε, σταθούμε σε αυτό που βρίσκω εμβληματικό και το γνωρίζουμε όλοι εδώ ως Επιτροπή το γεγονός ότι αυτός ο τομέας φαίνεται να μην αναγνωρίζει τα προβλήματά του. Ε, το νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν εδώ είναι ότι ευτυχώς είχαμε ήδη την έκθεση της Επιτροπής ΕΚΟΝ που είναι καθήλυνα αρμόδια όπως σωστά ε, θυμήσατε η οποία ασχολείται με τις ε, δεν ασχολείται καν μάλλον, δεν καλύπτει καν το θέμα των ε, βιομηχανιών οπτικοακουστικών, ούτε καν στην αιτιολογική έκθεση. Εδώ λοιπόν ο πολιτικός στόχος που ελπίζω να ε, είναι κοινό για όλους τους συναδέλφους είναι με αυτή την ευκαιρία να κάνουμε ε, κατανοητό στους συναδέλφους της Επιτροπής ΕΚΟΝ δύο σημαντικά σημεία. Πρώτον, την ιδιαίτερη διτή αξία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικροεπιχειρήσεων που γνωρίζουμε ότι είναι τόσο πολλές σε αυτό τον τομέα στα πολιτιστικά και τον τομέα της δημιουργίας. Είναι σημαντικό όχι μόνο για τον πραγματικό τους αντίκτυπο, για τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση αλλά και για τον ρόλο κλειδί που έχουν στην πρόθεση και την ενίσχυση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας Ως προς το δεύτερο αυτό σημείο, το είδος αυτός ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν δυσκολίες λίγο ακριβώς της δικής τους ε, οργάνωσης, των ιδιαίτερων ε, χαρακτηριστικών τους, λόγω της έλλειψης υλικών πόρων, την δυσκολία πρόσβαση σε άλλους πόρους, που κατ' επέκταση οδηγούν σε έλλειψη εγγυήσεων Κάτι που τους δυσκολεύει στο να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες και πιστώσεις. Επειδή υπάρχει περιορισμός βεβαίω στην έκταση της έκθεση που μπορούσαμε να συντάξουμε, θα δείτε ότι η έκθεση εδώ ε, έχει περισσότερο χρησιμοποιήσει μια γλώσσα στεγνή και κατανοητή. Κάτι που είναι περισσότερο μέρος των χαρακτηριστικών των της, ε, εκθέσεων τη Επιτροπή ΕΚΟΝ και όχι της δικής μας αλλά θέλουμε να συμπεριληφθούν τα σημεία που εμεί επισημαίνουμε στην τελική έκθεση τη ΕΚΟΝ. Θέλω να ολοκληρώσω ευχαριστώντα τη γραμματεία, ε, του συνεργάτε τη γραμματεία, κυρίω την δόκτωρα Φρανκ, για την πολύτιμη βοήθειά τη. Και μερικέ διευκρινήσει σε σχέση με το κείμενο. Ο στόχος μας είναι να δείξουμε με την έκθεση το ιδιαίτερο βάρος αυτού του τομέα και το πώς επηρεάζει συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Για το λόγο αυτό χρησιμοποίησα αριθμούς και στοιχεία της Eurostat. Να τα απαριθμίσω. Το 2014 τα άτομα που απασχολούνται στον πολιτιστικό τομέα ήταν 2,9 του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή 6,3 εκατομμύρια άτομα ποσοστό αυτό, το οποίο αξίζει να το πούμε, μπορεί να συγκριθεί με το εργατικό δυναμικό που αποσχολείται συνολικά στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα. Τη σύγκριση αυτή ήδη από, το, από την τάξη μεγεθών ελπίζω να καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να επηρεάσει και την Επιτροπή ΕΚΟΝ στη σύνταξη της έκθεσης αυτής. Αλλά γενικότερα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε, να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Οι θέσει εργασία στον πολιτιστικό και τον τομέα και τον τομέα τη δημιουργία μπορούν να χαρακτηριστούν ω ιδιαίτερες κοινωνικές προστιθέμενη αξία. Να τονίσω ότι συχνά οι θέσει αυτέ έχουν να κάνουν με ιδιαίτερε αρμοδιότητε και ανάγκε, πολιτιστικέ και ιστορικέ, που μπορεί να έχουν με τι ιδιαίτερε ανάγκε των περιφερειών και των επαρχιών. Και έχουν και άλλο ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι οι δύσκολα αλλάζουν χώρο. Επίση, ιδιαίτερη έμφαση στην έκθεση αυτή πρέπει να δοθεί στην ανάγκη να βελτιωθεί πρόσβαση στην πίστοση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει και τις μικροεπιχειρήσεις και να καλλιεργηθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες για την ορθή αξιολόγηση των ε, ε, εμπλεκομένων κινδύνων σε δύο μέτωπα. Πρώτα απ' όλα του κόστου που πρέπει να καλύψουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι δεν είναι τόσο έτοιμε να αντιμετωπίσουν τι απαιτήσει του τομέα του λογιστικού και των τραπεζών και μετά τι απαιτήσει των τραπεζών. Θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση στι πιστώσει για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, διότι αυτό είναι παραδοσιακό τρόπο χρηματοδότηση για τον τομέα τη ε, παρασκευή προϊόντων, τον ε, κλασικό τομέα. Αυτοί έτσι κι αλλιώ χρηματοδοτούνται εύκολα, αλλά οι τράπεζε, οι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν γνωρίζουν καλά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικροεπιχειρήσεων που ενεργοποιούνται στον τομέα αυτά. αυτό. Σε αυτό το τελευταίο παράδειγμα πρέπει να πω ότι όπως ε, μας λένε και οι μελέτες του ΑΣΕ πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συνολική αξιολόγηση κινδύνου και τη δυνατότητα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να γίνουν ενδεχομένω δεκτά ως εγγύηση για την παροχή δανείου. Έτσι μπορούμε να διευκολύνουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει με καινοτόμα συστήματα χρηματοδότηση, όπω τι μικρομε... μικροπιστώσει, το κεφάλαιο κινδύνου, το venture capital και ούτω καθεξής. Δεν θα σα πω τώρα όλε τι διαδικασίε. Άλλο σημείο που μπορούμε εδώ να υπογραμμίσουμε η ικανοποίηση από τον μηχανισμό εγγύησης στην δημιουργική Ευρώπη είναι ένας από τους τρόπους για να δοθεί μεγαλύτερη πρόσβαση στην πίστοση του τομέα αυτού της δημιουργίας και των πολιτιστικών διότι πραγματικά περιμένουμε ένα δις ευρώ το χρόνο απόδοση από το πρόγραμμα, από το εργαλείο αυτό βάσει των στοιχείων που έχουμε συγκεντρώσει ως τώρα και μας έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα την συλλογιστική αυτή να τη συμπληρώσουμε και φαντάζομαι οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν με μια τροπολογία. Μια τροπολογία που θα λέει ότι το ποσό αυτό πρέπει να ε, συμπληρωθεί και να εντοπίσουμε ένα χρηματοπιστωτικό κενό που αφορά και τις χαμένες επενδύσεις στην περίπτωση των επιχειρήσεων με ε, συγκεκριμένη εμπορική πολιτική ή ε, διαφορετικό προφίλ κινδύνου που τελικά δεν παίρνουν πίστοση ή μπορεί να μην υποβάλουν καν αίτηση διότι θεωρούν δεν έχουν αρκετά στοιχεία στον ηχητικό τους για να μπορέσουν να λάβουν ενίσχυση. Αυτά ήθελα να εντοπίσω και ελπίζω οι σκιώδεις εισηγητές να σημειώσουν με προσοχή τι παρατηρήσει μου και να παρέμβουν για να σχολιάσουν καθώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι οποίοι ξέρω ότι έχουν ιδιαίτερη αφοσίωση στο θέμα αυτό. Ο Τζαμπάτσκι. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το σχέδιο γλωμοδότησης. Το κείμενο είναι γεμάτο με τις συστάσεις της Επιτροπής μας όσον αφορά τον, την δημιουργική και πολιτισμική βιομηχανία. Καθώς ο Καλλιτεχνικό και δημιουργικός τομέας είναι μια μεγάλη, ένας μεγάλος τομέας. Πρέπει να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Εργάζομαι ως μέλος της Επιτροπής Τοπικών Υποθέσεων και σε διάφορες εκθέσεις για τα, διανοητικά, για τα δικαιώματα διανοητικής περιουσίας. Έχω πιστεί πως οι καλλιτέχνες αξίζουν μια δίκαιη αμοιβή πολλοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα δεν είναι μεγάλες επιχειρήσεις και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται χρηματοδότηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης προς εφαρμογή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Νέες ιδέες πρέπει να προσθεθούν στην γνωμοδότηση αυτή Μπορούμε να σκεφτούμε την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Horizon 2020. Επίσης, εστιάζουμε στο εργαλείο κόσμη για την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να εστιάσουμε αποκλειστικά στον, στην πολιτισμική και δημιουργική βιομηχανία. Ανεφ, κατέθεσα διάφορες τροπολογίες και ελπίζω πως τόσο ο συγκητής και οι άλλες πολιτικές ομάδες θα τις υποστηρίξουν. Η κυρία Evans. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πιστεύω πως έθεσε κάποια σημαντικά ζητήματα, τα οποία και παρουσίασε πολύ ωραία. Μου άρεσε ιδιαίτερα η σύγκριση μεταξύ των αριθμών των απασχολούμενων στην δημιουργική βιομηχανία με τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα Γνωρίζουμε φυσικά πως γενικά είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Γνωρίζω από την Ουαλία, όπου το 99% των επιχειρήσεων είναι μικροπεσές και η δημιουργία θέσεων εργασίας στον καλλιτεχνικό και δημιουργικό τομέα υπάρχουν διαφορές χρηματοδότησης τις οποίες και πρέπει να εξετάσουμε. Πιστεύω πως πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης πως εξετάζουμε κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη στα οποία γίνεται πολύ νομοθεσία, αλλά επίσης τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να υποστηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επειδή ο πολιτισμικός και δημιουργικός τομέας από τη φύση του αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της Ευρώπης, το οποίο είναι κάτι πολύ πολύτιμο. Επίσης θα ήθελα να επικροτήσω τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Πιστεύω πως αυτό έχει το δυναμικό ενός νέου συστήματος και αυτό θα ήθελα να, που θα ήθελα να θέσω ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το πρόγραμμα Δημιουργία Ευρώπη καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγοριοποιείται ως χώρα υψηλής παραγωγής, αυτό σημαίνει πως αιτήσει από οπουδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκλείονται από πρόσθετα μόρια, παραδείγματος χαρίως μειονεκτικέ συμπεριφοριακές περιοχές. Γι' αυτό και θα ήθελα να καταθέσω τροπολογίες σχετικά με αυτό συγκεκριμένα. Επειδή έχουμε δημιουργικότητα και δυναμικό, το οποίο ειστερεί για αυτόν τον λόγο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να κατατεθούν τροπολογίες αυτού του είδους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάμεμπερτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ο συνάδελφος Λουίτζι Μόργανο όντως έγραψε μια πολύ καλή γνωμοδότηση η οποία βάζει το δάχτυλο στην πληγή. Έχουμε μιλήσει συχνά γι' αυτό, το έχουμε διαπιστώσει συχνά επίσης. Ποιε είναι οι δυνατότητε τη χρηματοδότηση. Μιλήσαμε για την έλλειψη ειδικευμένη γνώση από τι τράπεζε για την αξιολόγηση κινδύνου. Και επίση το ερώτημα πώ μπορούμε στο μέλλον να διαμορφώσουμε καλύτερα το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Του χρόνου έχουμε τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, όπου πιστεύω πως μπορούμε να ξοδέψουμε κάποιες σκέψεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το πρόγραμμα αυτό στο σύνολό του. Όχι τόσο όσον αφορά τα οικονομικά, αλλά ίσως όσον αφορά τα θεματικά επίκεντρα. Και όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος, πιστεύω πως υπάρχει μια σειρά δυσκολιών. Επίσης όσον αφορά την, τον χειρισμό του, προγρι, του προγράμματος και την ευκολία των αιτήσεων. Πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό, αλλά είχα και μια άλλη σκέψη την οποία θα ήθελα να θέσω. στο πλαίσιο των τελευταίων διαβουλεύσεων σχετικά με τον μεσοπρόθεσμο χρηματοδοτικό σχεδιασμό αποφασίσαμε την προώθηση της, της πολιτισμικής οικονομίας να μην γίνεται μόνο από τη δημιουργική Ευρώπη, αλλά να πραγματοποιηθεί επίσης η δυνατότητα μέσω των διαφορετικών ταμείων να διατεθούν κονδύλια. Έχω ότι την εντύπωση πως τα διαφορετικά ταμεία βρίσκονται επίσης στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και οι δυνατότητες στα κράτη-μέλη είτε δεν είναι επαρκώς γνωστές ή τουλάχιστον δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς για να ζητηθεί και εδώ η προώθηση της πολιτισμικής και δημιουργικής οικονομίας. Επειδή υπάρχουν σαφώς περισσότερα χρήματα εκεί από ότι στη δημιουργική Ευρώπη. Γι' αυτό και πιστεύω πως θα ήταν μια καλή ιδέα εν συμπληρώναμε την έκθεση αυτή ως προς το ότι να προτρέπαμε επίσης την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχουν τα διαφορετικά τομεία για την χρηματοδότηση της δημιουργικής και της πολιτισμικής οικονομίας και να γνωστοποιηθεί αυτό, ότι έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια αυτά. Αυτή είναι μια πρόταση συμπλήρωσης που έχω, επειδή πιστεύω πως πρόκειται για μια σημαντική πτυχή, καθώς έχουμε πολύ περισσότερα κονδύλια εκεί από ό,τι στα μικρά προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε θέλει να μιλήσει κάποιος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλημέρα σας. Ραλούκα Πέιντερ με λένε. Εργάζομαι στο ε, γάμα δέλτα της Κομισιόν ε, για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίε και την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω σήμερα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί ε, στη δέκα του προηγούμενου έτου σε μια ευρεία διαβούλευση για τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για καλύτερη πρόσβαση ε, των ε, επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Γενικά μιλάμε για τις εταιρείες αλλά και ειδικότερα στις, ε, για τις ΜΜΕ και για τις νεοσυσταθήσεις εταιρείες, τις startups. Είχαμε λοιπόν αυτή την ευρεία διαβούλευση και πολλές συζητήσεις. Είχαμε και ένα συνέδριο εδώ στις Βρυξέλλες και μετά από όλα αυτά η Επιτροπή ενέκρινε το Σεπτέμβρη πέρυσι ένα σχέδιο δράσης. Δηλαδή έναν οδικό χάρτη με μια δέσμη 33 μέτρων που θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουν εφαρμοστεί μέχρι το 2019 προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εταιριών στη χρηματοδότηση. Και αυτός είναι ο ένας βασικός στόχος. Ένας άλλος βασικός στόχος είναι η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Αυτό μπορεί να γίνει με τα κεφάλαια πνευματικού κινδύνου business angels άλλες δηλαδή πηγές, όχι τράπεζες. Και το crowdfunding επίσης. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι στηρίζουμε και την ανάπτυξη οικονομικών ε, που βασίζονται στην αγορά για συμπλήρωση της δανειδότητας από τις τράπεζες, διότι οι μικρότερες επιχειρήσεις ε, θα συνεχίσουν να βασίζονται κυρίως ε, στα δάνεια από τις τράπεζες, αλλά αυτό το σχέδιο δράση τέλο πάντων θα πρέπει να θεωρηθεί ως ε, συμπληρωματικό και προς την υποστήριξη της ε, δανειοδότησης από τράπεζε. Για το θέμα αυτό συγκεκριμένα δε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι ζήτησε τη γνώμη των ενδιαφερομένων φορέων σε σχέση με τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία υλοποιήθηκαν μετά την χρηματοπιστωτική κρίση, ποιε είναι οι κεφαλαίκε τις τράπεζες και τα λοιπά και πώς όλα αυτά επηρεάζουν τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν τις ΜΜΕ. Τώρα είμαστε στην φάση που εξετάζουμε τι συνέχεια θα δώσουμε σε αυτή τη διαβούλευση για να δούμε ίσως ποια στοχευμένα μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για να διευκολύνουν, διευκολύνουν συγγνώμη, τις μικρότερες τράπεζες να μπορούν να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις μεταξύ των μέτρων τα οποία προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, συγκαταλέγεται ένας τομέας στον οποίο θέλουμε να εστιάσουμε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Τι εννοώ με αυτό, οι ΜΜΕ, πώς μπορούν να ενημερώνονται για αναλλακτικέ πηγές χρηματοδότησης αντί των τραπεζών. Συζητούμε λοιπόν αυτό τον καιρό με την, με την Ένωση των Τραπεζών και τις ε, ενώσεις ε, επιχειρηματιών για να δούμε κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία αφενό μεταξύ των τραπεζών και αφετέρου μεταξύ των ΜΜΕ. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα μια τράπεζα αρνείται να χορηγήσει ένα δάνειο, θα μπορούσε να ενημερώσει μια εταιρεία για το τι άλλε πηγέ χρηματοδότηση είναι διαθέσιμε. Αυτή είναι μια οδό. Μια άλλη οδό θα ήταν να γίνει μια χαρτογράφηση των συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμε σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διότι γνωρίζουμε ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν τέτοιε υπηρεσίε και είναι χρήσιμε για τι επιχειρήσει. Προσπαθούμε επίση να προωθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, σε ευρύτερη κλίμακα και μέσω μακροπρόθεσμα να δούμε πού υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας όπου θα μπορούν ε, οι ΜΜΕ να, να έχουν επαφή με τους επενδυτές. Να υπάρχει δηλαδή μια διαδικτύωση επενδυτών ε, και εταιριών που αναζητούν χρηματοδότηση. Επίσης τα venture capital, έχουμε την αθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ε, και έχουμε και τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ταμείου που θα προσελκύει δημόσιες και θετικέ επενδύσεις. Θα είναι ένα ταμείο λοιπόν μεγαλύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να στηρίξει ε, την παροχή κεφαλαίων. Μέχρι τα τέλη του μήνα μάλλον θα έχουμε γκρίνει και μια έκθεση για την κατάσταση ε, με την συλλογή κεφαλαίων, το crowdfunding και από νομοθετικής πλευράς να δούμε ποιοι ε, νόμοι έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο και πώς μπορούμε να στηρίξουμε την του crowdfunding προστατεύοντας ταυτόχρονα τους επενδυτές. Κάτι άλλο που θέλουμε να δούμε είναι και το βαθμό, το εύρος των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και πώς μπορούμε να στηρίξουμε την ασφαλή περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του μέσου χρηματοδότησης. Όπως είπα, υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία αποσκοπούν σε δημιουργία ενός α, πιο, πιο φιλοεπιχειρηματικού περιβάλλοντος σε, σε κάποιες χώρες. εστιάζουμε σε κάποιες διαδικασίες, ιδίως ε, στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και έχουμε τώρα ε, μια διαβούλευση ε, που γίνεται σε επίπεδο της ΓΔ δικαιοσύνη, DG Justice, που ίσως προτείνει και μέχρι τα τέλη της χρονιάς μια νομοθεσία περί μιας ελάχιστης εναρμόνισης στον τομέα αυτό. Στόχος μας λοιπόν όπως είπα είναι και η ενίσχυση, υποστήριξη αλλά και διαφοροποίηση, παροχή δηλαδή περισσότερων επιλογών για τις επιχειρήσεις. Ιδίω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω... Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο και όλους όσοι θα στείλουν τροπολογίες. Νομίζω όλοι συμφωνούμε να επικεντρωθούμε στην έκθεση αυτή, στην πρόσβαση στην πίστοση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ποικιλομορφία των πηγών χρηματοδότησης στην Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Νομίζω ότι αυτό ήταν ε, η ουσία όλων των παρεμβάσεων και υπό το φως αυτών θα υποβάλουμε μια έκθεση συνολική που θα ακολουθεί την κατεύθυνση που αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερη σημασία για την Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό βάρος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείε των τομέα των πολιτιστικών και, ε, πολιτισ, και ε, ε, για να συμπεριληφθούν και στην κοινή έκθεση ιδέε πρωτοβουλία τη Επιτροπή ε, που είναι καθήλυνα αρμόδια και θα αποβληθεί στι αρχέ καλοκαιριού. Ελπίζω ότι με του τροπολογίε θα βρούμε και τι απαραίτητε συμβαστικέ λύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φτάσαμε στο επόμενο σημείο. Στα διάφορα έχετε να πείτε τίποτα, τότε απλώς να σας πω ότι θα ξανασυναντηθούμε στις 25 Απριλίου, Δευτέρα στις 3 και εκεί θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας όπως και στις 26 Απριλίου στις 9. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την ε, η δεύτερη αυτή ημέρα συνεδρίασης, ευχαριστώ και τους διερμηνείς, καλή σας ημέρα.